Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να συμπεράνω ότι μπορεί να χάσουμε αυτή τη μάχη, αλλά δεν σημαίνει ότι χάσαμε και τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Εάν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σας κάνω μία ανακοίνωση. Θα ήθελα να πω ότι στις 9 Μαρτίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, εξέφρασε, μάλλον ε, υπερψήφισε ένα ψήφισμα σε σχέση με την ανισχυτική κατάσταση στη Σρι Λάνκα και σε αυτή την σύνοδο δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού ε, λήφθη υπόψη αυτή η πρόταση. Δηλαδή πριν από τις 12, ε, αν πριν από τις 12 αύριο το μεσημέρι 40 βουλευτές ε, ε, το ζητήσουν, τότε θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία. Μετά από αυτή την ανακοίνωση ας ξαναφτάσουμε στον ήρμό μας, στο μύτο της συζήτησης. Το λόγο έχει η κυρία Τσικάου, εξ ονόματος των ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ελκαντράουη και τον κύριο Γερζεμπόφσκι